του Κοινοβουλίου μας. Έλαβα από τις ομάδες ALDE και ENF κάποια αιτήματα διορισμού στις αντιπροσωπείες τους. Οι διορισμοί αυτοί θα καταγραφούν στα πρακτικά της τρέχουσας συνόδου. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών, οι διορισμοί αυτοί θα θεωρηθούν έγκυροι.